Ας ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίαση. Πριν προχωρήσουμε στις προφορίες, να επαναλάβω τα χθεσινά τα συγχαρητήρια που έστειλα το πρωί για την ανάληψη καθηκόντων υπουργού που θα αναλάβει ο συνάδελφος από την Πολωνία. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλη την, ε, από όλη την Επιτροπή. Ο συνάδελφος Δαρκόφσκι μάλλον θέλει το λόγο και τον έχει. Πολύ σύντομα. Να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε. Ήταν πραγματική μου χαρά να εργαστώ κάτω υπό την ηγεσία σας και μεγάλη μου χαρά να εργαστώ στην Επιτροπή ΑΦΚΟ με όλους σας. Ήταν μια σημαντική εμπειρία. Συνήθως όσοι αναλαμβάνουν ε, καθήκοντα υπουργού, ακόμη και αν έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο, είναι πολύ χαρούμενοι. Θα μου λείψετε όμως πολύ. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς να καταλάβει πώς μπορεί να λείψει σε κάποιον η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά για μένα αυτό ισχύει. Θα είμαι βέβαια εδώ στις 3 Δεκεμβρίου επισήμως, ε, θα είμαι μέλος. Οπότε για ό,τι χρειαστείτε θα είμαι στη διάθεσή σας. Μετά από αυτή την ημερομηνία θα προσπαθήσω να είμαι σε επαφή με το Ευρωκοινοβούλιο. Ίσως όχι για συνταγματικές υποθέσεις, διότι δεν θα μπορώ να ασχολούμαι πλέον με αυτά τα θέματα, αλλά θα είμαι υπεύθυνο για την ψηφιακή οικονομία και την δίκηση. Οπότε, ίσως Εάν δεν τα καταφέρω με την ε, προάσπιση του ψηφιακού μας συστήματος και συμβεί το παραμικρό, μπορεί να απολυθώ και να με ξαναδείτε εδώ. Αλλά ελπίζω όχι στην ερχόμενη πενταετία. Δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ παρά ως κάποιος που παρίσταται στις ακροάσεις σας. Πάντως σας ευχαριστώ γιατί αυτό που πέτυχα πλέον το χρωστάω σε μεγάλο μέρος εσάς. Ευχαριστώ. Και εμείς κυρία Υπουργέ και εμείς ε, πολεμήσαμε με αντίθετα συναισθήματα. Από τη μια φορά την, ε, είχαμε δυσάστα συναισθήματα γιατί πάντα συνεισφέρατε στις εργασίες επιτροπής. Από την άλλη είχαμε και τη χαρά διότι είδαμε ένα φίλο ένα ε, ιδιαίτερα πρικισμένο άτομο που αγαπάει την Ευρώπη να είναι μέλος της πολωνικής κυβερνήσεως. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη. Ψηφίζουμε την έκθεση Ταρκόρσκι. Λοιπόν, όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης και αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν ψηφίζουμε αυτές που συμπεριλαμβάνονται οι 4, 2, δύο τμήματα, 1, 12, 15, Τροπολογία 14, 13 και ακόλουθε. καταπίπτουν διότι είναι σε αντίθεση με τη σημαστική. Πάμε στην τροπολογία Β του συγητού υπέρ. Θα τα πείτε κάτι. Ορίστε. Είχα προτείνει σημαντική Α, Β και Δ. Εκεί είχα προτείνει προφορική τροπολογία και δεν ζητήσατε. Θέλω, θέλω τώρα να αναφέρω την προφορική τροπολογία, να εξηγήσω αν και ψηφίστηκε η Α. Τι τροποποίησα. να συμπεριληφθούν οι διεθνεί συνθήκε που δεν αντικατοπτρίζονται από τη συμβαστική και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αυτέ οι λέξει. Διεθνεί συμφωνίε στι συμβαστικέ. Διότι αν θυμόσαστε, το όλο θέμα για το άρθρο 81 είναι να αντικατοπτρίζεται η περίπλοκη κατάσταση που αφορά τις διεθνείς συμφωνίες. Και θα έλεγα ότι πρέπει να συμπεριληφθούν αυτές οι λέξεις στο, στο κείμενο. Ο κ. Σταρκόφσκι, με κάθε σεβασμό διαφωνώ. Η όλη ιδέα ήταν να συζητήσουμε το 81 και θα πιστέψουμε στην έκθεση όταν πάμε στο 90 άρθρο 95, παράγραφος 5, διευκρινίζει τη σύμφωνη γνώμη που έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σύμφωνες νόμους. Το συζητήσαμε επί μακρόν στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Θέλαμε να κάνουμε διάκριση και διευκρίνηση μεταξύ 81 και 90 και επενθυμίζω ότι εξακολουθούμε την επεξεργασία του άρθρου 90 που αφορά τις διεθνείς ε, συμφωνίες. Ψηφίσαμε τη συμβαστική Α και ας πάμε στη συμβαστική Β. Απλώς αυτό. Ο Πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Κατανοώ τη θέση, λέει ο κύριος Σόλτς, να ψηφίσουμε τότε τι τροπολογίες 15, 16 και 23 ξεχωριστά, διότι η εμπειρία από τις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες και από την Επιτροπή Ίντρα έχω αυτή την εμπειρία ότι χρειαζόμαστε τώρα αυτή τη διευκρίνηση. Είμαστε στη φάση διεθνών συμφωνιών που και γι' αυτό θέλω για τη 15, τη 16 και την 23 ξεχωριστές ε, ψηφοφορίες. Θεωρώ ότι στην πραγματικότητα αυτές η, αυτή Αυτροπολογία προφορική επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Ήδη στο άρθρο 90 αναφέρει στη πέμπτη παράγραφο ότι στην αρχή των διαπραγματεύσεων πριν την υπογραφή της συμφωνίας, κάθε συμφωνία στο σχέδιο συμφωνίας υπόκειται υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση για έγκριση. Η διαδικασία της έγκρισης πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 81. Είναι, ήδη υπάρχει αναφορά στο άρθρο 81. Δεν έχω πρόβλημα να το ψηφίσουμε, αλλά νομίζω ότι είναι άχρηστο, περιττό. Θεωρούσα ότι η σιωπή από αυτού του σημείου ε, θεωρεί το ως σύμφωνη γνώμη ή απόσυρση. Αν επιμένετε να ψηφίσουμε τις επόμενες συμβαστικές. Καλώς. Φτάσαμε στη συμβαστική Β λοιπόν. Υπέρ Σηκώστε το χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα, καλύπτονται τροπολογίες 1, πρώτο και δεύτερο τμήμα, 6, 5, 12, 28, 16, Σόλτ 16. Κύριε Σόλτ, θέλετε να ψηφίσουμε το 16. Εντάξει, ψηφίζουμε την τροπολογία 16 Σόλτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα δεν ψηφίζουμε ότι καλύπτονται την 24, τη 18, τη 12, τη 19, 17. 19. Σόλτς πρέπει να ψηφιστεί υπέρ της τροπολογίας 19, σηκώ στο χέρι. Κατά. Απορρίπτεται. ψηφίσαμε τη συμβαστική C, στη συμβαστική D πάμε τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα δεν ψηφίζουμε όλες τις τροπολογίες που καλύπτονται. Πάμε στο πρώτο τμήμα της τροπολογίας 1. Στην τροπολογία 1. Άρθρο 81 παράγραφος 2. Ζητώ συγγνώμη αν εφαρώ το σημείωμά μου. Και αυτό καλύπτεται στη συμβιβαστική. Μπορούμε να πάμε στην ε, συμβαστική. Υπέρ της ε κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία σχετικά αφορά την πρόταση αποφάσεως υπέρ, λένε ότι άρθρο 81 παράγραφος 2 πέμπτο τμήμα η τροπολογία του συγγητού πρέπει να ψηφιστεί. Πρέπει να ψηφιστεί. Σαφές. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 1 πέμπτο τμήμα του εισηγητού. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία υπέρ της προτάσεως κατά άποχες εγκρίνεται 16 υπέρ καμία ψήφος εναντίον, μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στον συγκητή, τον κύριο Ταρκόσκη. Είναι η τελευταία έκθεση που συζητούμε εδώ μαζί, μαζί σας, έτσι. Ψηφίζουμε λοιπόν το άλλο θέμα. Σχέδιο γνωμοδότησης για την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάλι Ταρκόσκι. Μέσορ Σμιτ μάλλον. Ο κ. Μέσορ Σμιτ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Δυνάτος το χειρός, παρακαλώ. Θέλετε να μιλήσετε. Ο κ. Μέσορ Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να ζητήσω συγγνώμη προς τα μέλη της Επιτροπής για κάποια θέματα διοργάνωσης. Δεν πήγαν πολύ καλά χθε. Συμφώνησα να έχει αποσταλεί εγκαίρω στους συναδέλφους η έκθεση ώστε να μπορέσει να ψηφιστεί σήμερα. Κάτι δεν πήγε καλά, αλλά παρόλα αυτά νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Το έχουμε ήδη συζητήσει μια φορά. Η γενική εντύπωση είναι ότι υπάρχει συνένεση για την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη-μέλη και για όσους ε, δεν ε, συμμορφώνονται υπάρχει μηχανισμός ε, επιβολής της οδηγίας και ελέγχου. Δεν φάνηκε χθε κάποιο να έχει κάποια αντίρρηση, οπότε, ούτε από τι τροπολογίε. Οπότε ελπίζω η ψηφοφορία να μπορεί να διεξαχθεί ομαλώ. Ακριβώ. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε και στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Διανάταση στις κύριες, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Χέφνερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Νταφ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κανείς εγκρίνεται. Μία ψήφο κατά καμία εποχή. Ε, απομένει η γνωμοδότηση που αναφέρεται και στην εμείς διάταξη για το άρθρο 302 για το άρθρο 202, μάλλον παράγραφος 5 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οργάνωση εξεταστικών αποστολών. Τα έχετε και στα ντοσιέ σα. Φαντάζομαι ότι έχετε το χρόνο να το δείτε. Υπέρ λοιπόν κατά αποχές εγκρίνεται με 17 ψήφους υπέρ, καμία κατά και καμία αποχή. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες, μπορούμε να επιστρέψουμε στην εμμυρίσια διάταξη. abbiamo siamo arrivati se non erro al punto Εάν δεν σφάλω, έχουμε φτάσει στο σημείο 15. καθεστώς και χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Ah, sì, c'era da vedere. Allora, sono Δύο σημεία μας έμειναν γιατί δεν είδαμε χθε την τροποποίηση του άρθρου 136 του κανονισμού σχετικά με τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδριάσεις. Και μεταμένει και αυτό των πολιτικών κομμάτων, όμως η εισηγήτρια δεν είναι στην αίθουσα. Θα μπορούσα βέβαια εγώ να την ε, αντικαταστήσω και να σας ενημερώσω για τα όσα συμβαίνουν, ενώ για το θέμα του 136 ο εισηγητής Χέφνερ, πού είναι ο Χέφνερ, ο Χέφνερ να πάρει το λόγο για το σημείο αυτό. Έπρεπε να το έχουμε δει από χθε, αλλά μας έμεινε, από... μας έμεινε για σήμερα, επειδή χθε είχαμε... δεν ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι είναι επίμαχο το θέμα, ούτε διαφέρουν πολύ οι θέσεις μας. Πρόκειται για μια μικρή έκθεση για τις υποθέσεις του Κοινοβουλίου. Θα θυμάστε ότι πριν από έξι μήνες περίπου λάβαμε μια επιστολή ε, η πρωτοβουλία ήταν της συναδέλφου Φραντσίσκα Μπραντνερ και υπέγραφαν και 25 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήθελαν στα πρακτικά των ε, συνεδριάσεων των επιτροπών να προσθεθεί μια καινούργια κατηγορία. Κατηγορία για τα μέλη που είναι σε άδεια μητρότητας ή πατρότητας, διότι οι άδειες αυτές, μητρότητας και πατρότητας, νομικά ε, μπορούν να δοθούν σε όλους και όποιος ασκεί την άδεια, τη χρησιμοποιεί, τη, ε, παρουσιάζεται ως αδικαιολογήτος απόν στα πρακτικά των συνεδριάσεων ε, και οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι που αξίζουν συγχαρητήρια αφού έγιναν πατέρες και μητέρες ε, παίρνουν ειδοποιήσεις ότι παραμελούν τις τα κοινοβουλευτικά τους ε, καθήκοντα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι και άλλες ομάδες ε, που κοινοποιούν τις λίστες των απόντων και κάνουν τους υπολογισμούς τους και έτσι φτιάχνουν, αν θέλετε, μια έκθεση για το εργασιακό ήθος των ε, βουλευτών. Μια έκθεση η οποία αξιώνει ότι θέλει να ε, αντικατοπτρίζει το εργασιακό ήθος των βουλευτών. Ε, πράγμα που δεν είναι σωστό αν δεν διευκρινίζεται. Ε, έτσι λοιπόν εκλήθην να υποβάλω μια έκθεση και το κάνω ακολουθώντας το δρόμο που πρότειναν οι συνάδελφοι, δηλαδή στον κανονισμό να προσθεθεί μια διάταξη που θα λέει ότι σε περίπτωση απουσίας λόγω άδεια μητρότητας ή πατρότητας να μην καταγράφεται η απουσία στα πρακτικά. Αυτό όμως, αυτό νομίζω ότι είναι προβληματικό. Ούτε νομίζω ότι μπορούμε να ε, συμπεριλάβουμε μια διάταξη που θα περιλαμβάνει κριτήρια που θα παρεκκλίνουν από άλλα σημεία του κανονισμού. Ε, κριτήρια για δικαιολογημένες απουσίες Εμείς ξέρουμε τις δικαιολογημένες απουσίες, μπορεί κανείς ε, να ε, απευθυνθεί στον πρόεδρο και να ζητήσει συγγνώμη. Το θέμα ρυθμίζεται από τους κοσμήτορες στο άρθρο 31 των εφαρμοστικών διατάξεων. Και έτσι θα ρυθμιστεί και ένα άλλο θέμα, γιατί πολλοί συνάδελφοι ήλθαν και με βρήκαν και μου είπαν τι γίνεται όμως σε περίπτωση υιοθεσία αν το παιδί δεν είναι το δικό μου το παιδί μετά από φυσική ε, γέννηση αλλά πρέπει να πάρω κάποια άδεια για να μείνω με το παιδί, να ε, ε, εξοικειωθούμε, να γνωρίσουμε ένα τον άλλον ή αν έχω ένα υπηρεσιακό ταξίδι για λογαριασμό του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να εφευρίσκουμε καινούργιες κατηγορίες. Η πρόταση είναι στο άρθρο 31.4 του εφαρμοστικό κανονισμό ε, να τον ε, υιοθετήσουμε γιατί εκεί αναφέρεται η δικαιολογημένη απουσία. Μπορούμε λοιπόν να εντάξουμε στο άρθρο το δικό μας 136 μια διάταξη που θα λέει απλά ότι στις περιπτώσεις όπου οι βουλευτές λείπουν δικαιολογημένα να γράφεται στο, στα πρακτικά ως ε, χωριστή κατηγορία, δηλαδή να είναι οι παρόντες εκείνοι που με την υπογραφή τους ε, γράφονται στον κατάλογο των παρόντων και υπάρχει και η οι απόντες, οι δικαιολογημένα απόντες και μια τρίτη κατηγορία ε, μη αδικαιολογήτως απόντες. Αυτή είναι η πρόταση που δίνει τη δυνατότητα στους συναδέλφους να καταγράφεται τακτικά και νοικοκυρεμένα στα πρακτικά ε, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη νέων ε, διατάξεων στο ε, δικαίωμα μας και η απόφαση λαμβάνεται από τον Πρόεδρο βάσει των προτάσεων των κοσμητόρων. Προτείνω λοιπόν με βάση το άρθρο 212 να κάνουμε μια τροπολογία στο άρθρο 136 όπως σας το είπα ε, σύντομα και τακτικά που θα λύνει το πρόβλημα για όλους τους ενδιαφερομένους. Και περιμένουμε ενδιαφέρον τις αντιδράσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος το λόγο για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Thank you so much, Mr. Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα αυτό. Ο συνάδελφος κύριος Μάρτιν ήθελε να μιλήσει ε, για αυτό το θέμα, αλλά ασθενή και δεν μπόρεσε να έρθει στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, μου ζήτησε λοιπόν να μιλήσω εγώ. Το παράδοξο αυτής της υπόθεσης είναι ότι Μόλις επέστρεψα από άδεια μητρότητας, οπότε ε, θα έλεγα ότι δικαιούμαι να μιλήσω για το θέμα. Και είναι απόλυτα σωστό να αναγνωριστούν από το Κοινοβούλιο αυτές, αυτοί οι λόγοι απουσίας, όπως οι άδειε μητρότητας, πατρότητας για τα μέλη. Δεν είναι το ίδιο όπως απουσία. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Το δε Κοινοβούλιο θα πρέπει να δίνει το παράδειγμα ε, τονίζοντας ε, την σημασία των ε, αδειών λόγω πατρότητας και αμητρότητας και ασθενείας. Εγώ ερωτήθην πολύ από τα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της άδεια μητρότητας, πώς το ρυθμίζω δηλαδή και δεν μπορούσα να απαντήσω ικανοποιητικά για τα μέσα ενημέρωσης. Ενώ τώρα με την έκθεση αυτή οι διαδικαστικοί μας κανόνες θα αναφέρονται στα μέλη που δικαιολογούνται από τον πρόεδρο. Τώρα δηλαδή υπάρχουν πρόσθετη λόγοι απουσίας, δικαιολογημένης απουσίας και θα περιλαμβάνονται και στα εκτελεστικά μέτρα τα οποία χειρίζονται οι κοσμήτορες, οπότε είναι εντάξει αυτό. Το αρχικό αίτημα των βουλευτών που υπέβαλαν την πρόταση και την τροπολογία αναφέρονταν μόνο στις άδειες μητρότητας και πατρότητας. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας και άλλους λόγους όπως ασθένεια, να, όπως στην περίπτωση του συναδέλφου κυρίου Μάρτιν για παράδειγμα και κοινοβουλευτικό έργο αλλού. Η Επιτροπή πρέπει όμως να συζητήσει ακριβώς ποιοι λόγοι θα θεωρηθούν δικαιολογημένοι για την απουσία. Η επεξηγηματική έκθεση του εισηγητή, η αιτιολογική έκθεση, εξηγεί πάρα πολύ ωραία τους λόγους ε, για την τροπολογία, ε, ο κατάλογος των παρευρισκομένων είτε ευρέως, ε, κοινοποιείται σε πολλά πρόσωπα που παρευρίσκονται και καταγράφει τις τάσεις στην προσέλευση των βουλευτών στις συνεδριάσεις. Ε, το website VoteWatch αναφέρεται ειδικότερα στην θεολογική έκθεση γιατί χρησιμοποιείται από πολλούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως ε, δεν χρειάζεται να αναφέρομαι έναν ιστότοπο, να αναφερθούμε ειδικά στο VoteWatch, ε, αυτό θα το σκεφτεί ο εισηγητής αφού μόνο ο εισηγητής μπορεί να τροποποιήσει την αιτιολογική έκθεση. Γενικά, ο σκιώδης των σοσιαλιστών στηρίζει την έκθεση χωρίς άλλες προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, ναι, δεν έχω αντίρρηση, καμία αντίρρηση όσον αφορά την πρόταση. Όπως βλέπω τα πράγματα, ισχύει μόνο για την Ολομέλεια, διότι η παρουσία στις επιτροπές δεν κάλυπτεται από την Vote Watch. Μπορεί να βρει κανεί τον αριθμό των παρουσιών στις επιτροπές, αλλά είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί. Μήπως μπορεί να αναφέρετε ρητά ότι δεν ισχύει αυτό μόνο για την παρουσία στην Ολομέλεια, αλλά επίσης και για την παρουσία στις Επιτροπές. Ε, Έλεγα λοιπόν, όσον αφορά τις επιτροπές ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να επεκτείνουμε την πρόταση του συναδέλφου Χέφνερ. Μπορούμε να κάνουμε τροπολογίες όμως. Μπορούμε να θέσουμε την προθεσμία υποβολή τροπολογιών 5η 12 Δεκεμβρίου το μεσημέρι η 12 δεκεμβριου το μεσημερι ψηφοφορια θα πρέπει να γίνει αν συμφωνήσει ηγητής στις 21 Ιανουαρίου. Αποφασίζεται ούτως. Θέλετε κύριε να πείτε κάτι. Όχι να πω πολύ σύντομα. Πρώτον ότι ρυθμίζονται όλες οι περιπτώσεις όπου βάσει του κανονισμού η παρουσία, η παρουσία κοινοποιείται. Δεύτερον, προφανώς όταν υπάρχει ε, να, να ε, αναφερθούμε γενικά σε ιστότοπους χωρίς το Vote Watch, να το κάνουμε και αυτό. Ε, και τέλος ε, υπάρχει μια μικρή αναγκαία τροποποίηση, γιατί νομίζω ότι δεν είναι σωστό οι συνάδελφοι στη σημερινή δημοκρατία των μέσων να εγκαλούνται για κάτι που δεν είναι μόνο δικαίωμά τους, αλλά και υποχρέωσή τους σήμερα ε, ε, στα πλαίσια του ρόλου τους ως γονείς. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αυτή την ε, τροποποίηση στον εσωτερικό κανονισμό και νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα ούτως ώστε ικανοποιητικά να επιληθεί το θέμα για τους συναδέλφους. Νομίζω ότι είναι θετική αυτοποθέτηση όσον αφορά την πρόταση. Δεν είναι κάτι πολύ κατεπήγον. Γι' αυτό εγώ έθεσα την προθεσμία για τις τροπολογίες 12 νομίζω Δεκεμβρίου. Μεσημέρι η ψηφοφορία θα γίνει στην Σύνοδο του Ιανουαρίου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο σημείο που αφορά το, τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, το σχετικό καθεστώ για τα ευρωπαϊκά κόμματα και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Η κυρία Γιαννάκου είναι η συγκήτρια. Δεν είναι παρούσα, αλλά συμφωνούμε, συμφωνήσαμε να σα δώσω εγώ τι πληροφορίε. Στι 19 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο Έγινε ο δεύτερος τριμερής άτυπος ε, διάλογος υπό Λουθανική Προεδρία και το άρθρο 70 του κανονισμού καθορίζει ότι μετά από κάθε τριμερή διάλογο η διαπραγματική ομάδα θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή και σε αυτή την περίπτωση εμάς. Ποιες πληροφορίες μπορώ να σας δώσω. 19 Νοεμβρίου λοιπόν, στον τριμερή διάλογο, ελπίζαμε το Συμβούλιο να έδινε συγκεκριμένη έντολη στην Λιθουανική Προεδρία. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα το Συμβούλιο ελείψη αναγκαίας πλειοψηφίας δεν ετοίμασε συγκεκριμένη έντολη. Έτσι, ο, η Λιθουανική Προεδρία, ο Πρόεδρος μπορεί σε συνοπτικό σημείο να διαβιβάσει και αναφέρει τα σημεία στα οποία το Συμβούλιο έχει πετύχει η συμφωνία. Ποια είναι τα σημεία. Η θέση του Συμβουλίου ποια είναι. Όσον αφορά τη διοικητική καταχώρηση, εγγραφή, πρέπει αυτό να γίνεται αυτόματα. Δηλαδή από τη στιγμή που πληρούνται οι τυπικές συνθήκες, οι τυπικοί όροι και γίνει η παλήθευση και υπάρχει γραπτή υποχρέωση ότι το κόμμα που ζητεί την, ε, να εγγραφεί θα σέβεται τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, τότε η καταχώρηση γίνεται αυτόματα, η εγγραφή. Συζητήσαμε επί μακρόν και αυτή τη φορά ποιος πρέπει να συμμετάσχει αυτή την εγγραφή. Εμείς λέγαμε ότι θα πρέπει το κοινοβούλιο να είναι το αρμόδιο όργανο στο οποίο θα γίνεται η καταγραφή που θα προβλέπει αυτή την υπηρεσία για την εγγραφή ενώ το Συμβούλιο πάντα υποστήριζε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτόνομη αρχή ο διευθυντή θα πρέπει να διορίζεται κατόπιν σύμφωνη γνώμη των τριών θεσμικών οργάνων, των ευρωπαϊκών, αλλά θα πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα. Το Συμβούλιο όσον αφορά τη διαγραφή έλεγε ότι αυτή η αρχή θα πρέπει να κάνει τη διαγραφή το, Συμβούλιο θα πρέπει, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και το Συμβούλιο να αντιταχθούν σε αυτή τη διαγραφή. Το καθεστώς των κομμάτων δεν έχει συγκεκριμένες ιδέες στο Συμβούλιο, δεν έχει κάνει προτάσεις. Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, η θέση του Συμβουλίου όπως κατεγράφει στις 19 Νοεμβρίου φαίνεται πως ανατελίζεται προς το να παραμείνει το status quo, να μην αλλάξει τίποτα. Το Συμβούλιο ε, πλησιάζει στη θέση του στην Διοργανική Συμφωνία. Δηλαδή για το θέμα της εγγραφής και διαγραφής και της αρχής, της αρμόδιας, όσον αφορά όμως τη χρηματοδότηση, το Συμβούλιο φρονεί ότι η χρηματοδότηση μπορεί να πάει στον υποψήφιο του Προέδρου, αλλά όχι στη χώρα. Η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου απάντησε με θέση διαφοροποιημένη για όλα τα σημεία. Στον τελευταίο άτυπο τριμερή διάλογο είπαμε ότι μπορούμε να υποχωρήσουμε όσον αφορά την εγγραφή, μπορούμε να δεχθούμε αυτή η εγγραφή του κόμματος να γίνεται από έναν φορέα ή μία αρχή, δεχόμαστε να είναι και νομικό πρόσωπο, και ο Διευθυντής να διορίζεται με την ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από φορέα του Κοινοβουλίου, Πρόεδρο ή άλλων, αλλά όσον αφορά τη διαγραφή δεχόμαστε τον αυτόματο χαρακτήρα τον αυτόματο χαρακτήρα και της εγγραφής, ονόματι της ελευθερίας, της έκφρασης, της σκέψης κλπ, της συγκρότησης ομάδας κλπ και τη συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα. Αυτό το δεχόμαστε. Όσον αφορά την διαγραφή από το αρχείο, είναι τόσο βαρύ αυτό, τόσο σημαντικό, σαν γεγονός από πολιτική σκοπιά, που θα πρέπει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορούν να τοποθετούνται από αυτού. Ο τελικός έλεγχος αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι μπορεί να γίνει προσφυγή, εν πάση περιπτώσει, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ίσως σε αυτήν την τελική φάση της διαγραφής πρέπει να υπάρξει συμφωνία, δηλαδή που θα λέει ότι η διαγραφή πραγματική γίνεται από την αρμόδια αρχή που κάνει και τις εγγραφές, αλλά αυτή η διαγραφή θα πρέπει να γίνεται μετά από ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και ενδεχομένω το Συμβούλιο. Εκείνο που αποφασίζει τελικά, σύμφωνα με τη θέση που εκφράσαμε εμεί, είναι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σίγουρα η αρχή αυτή αρμόδια της εγγραφή μπορεί να διαφωνεί επί της διαγραφής για λόγους τεχνικής φύσεω και νομικού λόγους, τότε ενδεχομένω με γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Σοφών θα μπορεί να απορριφθεί η διαγραφή, αλλά η διαγραφή όσον αφορά και την άρνηση της διαγραφής και τη διαγραφή, αυτό είναι κάτι που θα ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί βρίσκονται συζητήσει συζητήσεις λίγο πολύ. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία πολιτική στην διεκπαιρέωση αυτού του θέματος για τα πολιτικά κόμματα. Πιστεύω προσωπικά ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία και να πετύχουμε πάση θυσία συμβιβασμό βέβαια διατηρώντας τα βασικά στοιχεία των θέσεών μας. Το λέω αυτό διότι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι μας έδωσε σαν πρόταση, δεν το διάβασα ακόμα, ένα κείμενο, μια διατύπωση πιο ακριβή που αφορά ενδεχόμενη θέση που πλησιάζει πολύ τη θέση του Συμβουλίου κατά την άποψή μου και ζητά να γίνει άλλη άτυπη συνεδρία σε τεχνικό επίπεδο αυτή την εβδομάδα. Τίθεται το εξής ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν ένας τεχνικός τριμερής διάλογος που θα συμμετέχουν οι υπάλληλοι, εμπειρογνώμονες, μπορεί να προηγηθεί ή να ακολουθήσει τον πολιτικό τριμερή διάλογο, εκεί που αποφασίζονται οι κατευθύνσεις ο τριμερής τεχνικός διάλογος δίνει κάποια τάξη στις ε, πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την άποψή μου. Αλλά για να φτάσουμε γρήγορα σε διεκπαιρέωση του θέματος μας οδηγεί στο να συμφωνήσουμε και στη διεξαγωγή ενός τριμερούς ε, διαλόγου τεχνικής φύσης αυτήν την εβδομάδα. Επ' αυτού θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ε, ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Νταφ. Πρόεδρε, δεν είμαι βέβαιος ότι εκφράσατε ακριβώς τη θέση μας όπως το βλέπω εγώ. Νομίζω στο Συμβούλιο υπάρχει μια πλειοψηφία αρκετά μεγάλη υπέρ της πρότασης η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των τριών νομικών υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων. Τρία μόνον μέλη έχουν αντιρρήσει. στο Ηνωμένο Βασίλειο για προφανείς λόγους, οι κάτω χώρες, για λιγότερο προφανείς λόγους και οι Τσέχοι. που δεν έχουν κυβέρνηση. Νομίζω όμως ότι ο τελευταίος τρεμερής διάλογος ήταν ε, τελείως λιβερός με πολύ κακή διεξαγωγή της συζήτηση και η Προεδρία βρισκόταν σε τελείως, ε, σε πλήρη σύγχυση. Μιλάω για την Προεδρία του Συμβουλίου. Πέραν αυτού όμως και παρά τα αυτά υπάρχει ένα σχέδιο κειμένου το οποίο θα ήταν μια βάση από τις οποίες να μπορεί να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο. Δεν βλέπω το λόγο να οργανωθεί όμως ε, τριμερής διάλογος με τεχνικό περιεχόμενο χωρίς να συμβοληθούν τα πολιτικά ζητήματα. Κάτι που θα γίνει στην αρχή της επόμενης εβδομάδας και γι' αυτό βεβαίως χρειαζόμαστε το έγγραφα με τις τέσσερις στήλε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως, καταλαβαίνω εξ όσων μαθαίνω ότι ή το ετοιμάζουν ή τέλος πάντων κοντεύει να ολοκληρωθεί το κείμενο αυτό. Και δύο επί της ουσίας σημεία για το συμπεριεχόμενο του σχεδίου συμφωνίας. Το πρώτο, είναι για το άρθρο 12.4, εδάφιο 4. Θα πρέπει να παραμείνουν τα ποσοστά όσα έχουν και κατά δεύτερον για το θέμα που σωστά έγινατε κι εσείς για την οικονομική στήριξη υποψηφίου των επικεφαλής υποψηφίων που είναι υποψήφιοι και για το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να δούμε κατά πόσον το άρθρο που θα πρέπει να το επιλύει αυτό είναι το 18.1 και να δούμε κατά πόσον μπορεί να βρεθεί διατύπωση που να απαγορεύει την έμεση χρηματοδότηση υποψηφίων. Αλλά η διατύπωση για την άμεση χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει. Αυτό θα μπορούσε να άρει όλες τις νομικές επιφυλάξεις. Εγώ πρότεινα να συμφωνηθεί μια ταχεία διοργάνωση πολιτικού τριμερούς διαλόγου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Μπρόνς. Η αιτιολογική έκθεση λέει ότι μπορεί ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα να καταγραφεί αλλά να μην ζητήσει χρηματοδότηση. Αλλά δεν μπορεί να ζητήσει χρήματα χωρίς να έχει εγγραφεί. Πότε μπορεί να εγγράφεται αλλά να μην ζητάει χρηματοδότηση ένα κόμμα. Δεν βλέπω να υπάρχει νομική υποχρέωση εγγραφής και για το αίτημα για χρηματοδότηση Οπότε νομίζω ότι πιο εύκολο φαίνεται να ε, είναι το θέμα της εγγραφής παρά η εγγραφή συν η αίτηση για χρηματοδότηση. Τι μειονεκτήματα υπάρχουν από τη μη εγγραφή σε σχέση με την εγγραφή χωρίς όμως ε, απόκτηση χρηματοδότησης. Εσείς κύριε Πρόεδρε αναφερθήκατε στη διαδικασία της διαγραφής και είπατε ότι είναι σημαντικό πολιτικό θέμα. Η λέξη πολιτικό είναι καλά επιλεγμένη, γιατί παρόλο που μιλάμε για μεροληψία, η μόνη εφαρμογή που έγινε και αναφέρεται νομίζω στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι, ξεχνάει τη βάση επί της οποίας επιδιώκεται η διαγραφή που είναι ανάλογο με κάποιον που γράφει στην ε, αστυνομία και λέει ότι πρέπει κάποιος να διωχθεί και να φυλακιστεί χωρίς να αναφέρει το αδίκημα που διέπραξε. Το μνημόνιο, όπως και τα άλλα σχετικά έγγραφα, αναφέρεται στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, αλλά είναι ελευθερία του συνεταιρίζεσθε για τους εγκεκριμένους μόνο. Σταματώ επί του παρόντος εδώ, γιατί αυτά τα έχουμε ξαναπεί τόσες φορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ταρκόφσκι. Very briefly, uh... Πολύ σύντομα. Τα έχουμε πει πολλές φορές αλλά αν θέλουμε να κλείσει η συμφωνία και νομίζω ότι όλοι το θέλουμε αυτό να γίνει πριν από τις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις για τις προτεραιότητές μας. Η πρόταση όσο έχει τώρα επιτάπητος είναι αρκετά καλή, όχι τέλεια, αλλά καμιά φορά το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Το Συμβούλιο είναι λίγο αναστατωμένο Οπότε ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την Προεδρία και όλοι ξέρουμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη τη στηρίζουν, πιέζει περισσότερο εμάς. Μας ε, θέτει προ μεγαλύτερων ε, ευθυνών και προτεραιοτήτων που πρέπει να υπερασπιστούμε. Είναι σαφές ότι τα δύο-τρία θέματα που πρέπει να υπερασπιστούμε ε, πρέπει να κλείσουν και να κάνουμε συμβιβασμό να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Δεν μπορεί να ξαναφέρουμε όλα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Θα πρέπει να ε, περιορίσουμε τις ε, προτεραιότητες στη χρηματοδότηση και να επικεντρωθούμε στα δύο-τρία σημαντικά και να πιέσουμε μετά το Συμβούλιο. Μόνο έτσι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το φάκελο πριν από τις εκλογές. Αν συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή που δεν θα είναι αρκετά εστιασμένη, με αυτή την Προεδρία θα έχουμε πρόβλημα αν και όλοι ξέρουμε ότι και η Προεδρία δουλεύει σκληρά για να κλείσει ο φάκελος. Ας τους δώσουμε ένα χέρι λοιπόν, αλλά να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να υπάρξει πολιτική συμφωνία εδώ, σε μας. Και όπως είπα, ε, ένα ή δύο είναι τα πραγματικά προβλήματα όταν πρόκειται για την επαλήθευση και πρέπει να τα πούμε πολύ γρήγορα. Αυτά είναι τα εκρεμή ζητήματα, ε, γιατί αλλιώς θα κατακλειστούμε από λεπτομέρειες που εντάξει κάποιες μπορούν να βελτιωθούν αλλά στο τέλος δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία με αυτά και με αυτά. Λοιπόν, Χέφνερ και Σόλτς και μετά θα πω αυτά που θέλω εγώ. Κύριος Χέφνερ. Yes, I completely agree. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Πραγματικά πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αν υπάρχει καλή βούληση, μπορεί να βρεθεί λύση και γρήγορα. Έχει προετοιμαστεί αυτή η λύση. Εγώ ζήσα τη βοήθεια και είχα τη βοήθεια των νομικών υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων. Έχουμε κοινό έδαφος, έχουμε προτείνει λύσεις. Το σημαντικό κατά την άποψή μου είναι κάτι προφανές, ότι από πλευράς Κοινοβουλίου δεν είμαστε εκείνοι που επανειλημμένα θέτουμε τέτοια ζητήματα. Είμαστε ικανοποιημένοι με την επιτευχή σας συνένεση και θέλουμε να λύσουμε τα δύο-τρία εκρεμή ζητήματα. Προτείνω λοιπόν να διαλέξουμε επίσημο τριμερή διάλογο ή δυνατόν αυτή την εβδομάδα. Και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει αντιληπτό από τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη ότι θέλουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό και να καταλήξουμε σε λύση και συνένεση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο. Έχω την πεποίθηση ότι αν ο τριμερής αυτός διάλογος προχωρήσει σωστά, τον χειριστούμε σωστά, θα καταλήξουμε σε απόφαση. Και αυτή η απόφαση θα μπορέσει να στηριχθεί από το Συμβούλιο μετά τον τριμερή διάλογο. Προτείνω λοιπόν να ζητήσουμε επίσημο τριμερή διάλογο και να ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είχαν συμμετάσχει στον τελευταίο τριμερή διάλογο είναι κάπως απογοητευμένοι όσον αφορά την προθυμία του Συμβουλίου να προχωρήσει. Ο Άντριου Νταφ περιέγραψε την κατάσταση και συμφωνώ με αυτά που είπε. Προτείνω να προσπαθήσουμε να μπούμε σε επίσημο τριμερή διάλογο το ταχύτερο δυνατόν και να διατηρήσουμε την πίεση. Θέλουμε από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διεκπαιρεωθεί αυτό το θέμα. Αυτό είναι το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε. Αν επιμείνουμε σε αυτό το στόχο και αν προωθήσουμε τις θέσεις που προωθήσαμε μέσω των άλλων τριμερών διαλόγων, θα είμαστε θέση να πετύχουμε συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Υποστηρίζω όλους τους συναδέλφους που ζητούν επίσημο τριμερή διάλογο το ταχύτερο δυνατόν. Ε, io volevo ripetere... Κοιτάξτε, θα εκφράσω αυτή τη φορά καλύτερα την άποψή μου. Και εγώ είμαι αισιόδοξο. Στην ε, Επιτροπή μας και στη διαπραγματευτική ομάδα είναι σαφείς οι θέσεις. Ήδη καταφέραμε πολλά διότι η αρχική στάση ήταν εχθρική η, θέση κατά της Επιτροπής των Επευθύνων που θα λαμβάνει με ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα. Όμως αυτά που απομένουν ε, ερωτώ, ε, ως ανοιχτά ερωτήματα είναι σαφή πλέον αφού ξεπεράσαμε τους πρώτους κοπέλους. Μα τη χρηματοδότηση δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Τα θεσμικά ζητήματα. Ε, σε αυτά έχει γίνει ένα βήμα πρόοδου θα υπάρξει νομοθεσία, θα υπάρχει αυτόματη επίλυση του θέματος. Εδώ υπάρχει πιθανότητα σίγουρης ε, συμφωνίας. Τώρα, για την εγγραφή, Βεβαίω, ε, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν ένα κόμμα δεν είναι εγγεγραμμένο, δεν μπορεί να ζητήσει και χρηματοδότηση. Είναι σαφέ. Από τη δική μου τη σκοπιά, το μόνο πρόβλημα που απομένει από τη θεσμική πλευρά είναι το ένα και μόνο. Το θέμα της διαγραφής. Οι προτάσεις που έχω ακούσει στον τελευταίο άτυπο τριμερή λένε ότι θα πρέπει η αρχή εγγραφή να την αναλαμβάνει και αυτή τη εγγραφή. Εγώ το βρίσκω κάπως αντιφατικό για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η αποπομπή ενός κόμματος. Ε, ο αποκλεισμό του από τη ανταγωνισμού με τα άλλα κόμματα να είναι κάτι που θα το, θα αποφασίζει μια τέτοια επιτροπή. Ή τέλο πάντων κάποια υπηρεσία. Μου φαίνεται τελείω ε, αδιανόητο. Η συμβαστική λοιπόν για το σημείο αυτό θα μπορούσε να βρεθεί εάν σκεφτούμε τι γίνεται εάν ψηφίζει και το κοινοβούλιο σε αυτή την περίπτωση, αν γίνεται συζήτηση στο κοινοβούλιο. Διότι αν υπάρξει περίπτωση διαγραφής και θέλουμε να ισχύουν οι επίσημοι όροι που ισχύουν για την περίπτωση τη εγγραφή. Δηλαδή, σύμφωνη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, ότι θα πρέπει να φτάσει το ποσοστό του 3%. Όλα αυτά είναι επίσημη διαδικασία. Τότε, προφανώ, η αρχή εγγραφή μπορεί να διαπιστώσει κάποια πράγματα και να προτείνει την διαγραφή με απόφαση η οποία να, είναι, να μπορεί να αποβληθεί σε έφεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλά δεν μπορεί αυτό να το αποφασίζει ένα ε, μόνο πρόσωπο, ένα άτομο. Θα πρέπει να είναι απόφαση που να τη λαμβάνει το ύψιστο πολιτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και ω προ αυτό, και να ολοκληρώσω την σκέψη μου παρόλο που καταγράφω και τι δικέ σα, ε, θα ήμασταν κοντά σε μια λύση διότι η πρόταση όπως έχει έτσι συγκεκριμένα υποβληθεί από την Προεδρία της Λιθουανίας νομίζω δεν το έχω διαβάσει ακόμη το κείμενο, μου λένε όμως, μου λένε, έτσι έχω ακούσει. Δεν έχει υποβληθεί ακόμη επισήμως Η πρόταση προβλέπει την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν προβλέπει δευτερευόντως τι θα γίνει εφόσον ληφθεί απόφαση από την πολιτική αρχή. Ας πούμε λοιπόν ότι η πολιτική αρχή αποφασίζει τον αποκλεισμό και για λόγους περιεχομένου. Αλλά το κοινοβούλιο έχει αντίρρηση. Εμένα δεν μου φαίνεται ότι πρέπει να λειτουργεί έτσι αυτό ο μηχανισμό. Το Κοινοβούλιο και αν θέλει και το Συμβούλιο κατά την άποψή μου πρέπει να αποφασίζουν τον αποκλεισμό ενό κόμματο αλλά συνεπώς με όσα επισήμως προβλέπονται. Διαγραφή της εγγραφής. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει διαγραφή της εγγραφής η οποία ουσιαστικά ε, λαμβάνεται υπόψη και εκτελείται από την ε, αρμόδια αρχή. Την απόφαση της διαγραφής. Ποιος τη λαμβάνει. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να αναζητηθεί συμφωνία. Διότι αν στον ε, τεχνικό άτυπο τριμερή διάλογο πρέπει να τοποθετηθώ. Θα ακολουθήσω από την άποψή σα, αλλά ω προ αυτό θεωρώ ουσιαστικά ότι είναι απλώ θέμα διατύπωση. Οι νομικοί πυρογνώμονε μπορούν να υποβαλούν και μια εναλλακτική πρόταση. Δεν είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να είναι πολύ σαφώ καθορισμένο. Διότι στην πραγματικότητα η σύγχυση η οποία έχει διαφανεί και έχει προκληθεί σε όλους τους τριμερείς διαλόγους είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση εδώ. Ε, μιλάμε και διαφορετικέ γλώσσε, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώ ο ένα τι λέει ο άλλο. Θα πρέπει κάτι να το γράψουμε για να υπάρξει και μια σαφή επιλογή μεταξύ εναλλακτικών, ή τη μία ή την άλλη. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει παρέμβαση του Κοινοβουλίου για τη διαγραφή, εφόσον υπάρχει πρόβλημα με τι αξίε, αλλά δεν ξέρουμε πού να το βάλουμε αυτό το πράγμα. Πού να τη βάλουμε αυτή την παρέμβαση του Κοινοβουλίου άλλο η ηλική ε, εκτέλεση της διαγραφής. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει άλλο πολιτικό πρόβλημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Παρ' όλα αυτά είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω και τις δικές σας ιδέες και απόψεις. Ο κύριος Νταβ, κύρια Γκουρμά και ο κύριος Χέφνερ. Πρόεδρε, με κάθε σεβασμό νομίζω ότι δεν πρέπει να προσπαθείτε να περιπλέκεται περισσότερο τα πράγματα από ό,τι ήδη είναι. Στο κείμενο του άρθρου, στο σχέδιο κειμένου, για τη διαγραφή, είναι αρκετά σαφή τα πράγματα. Είτε το Κοινοβούλιο, είτε το Συμβούλιο δίνανται να αντιταχθούν στην απόφαση της αρχής περί διαγραφής ενός κόμματος. Είμαστε εμείς τελικά η θέση παναχώρησης. Εμείς είμαστε σε θέση να ελέγξουμε αυτή την απόφαση μάλλον. Αυτή η διατύπωση πλήρως καλύπτει τις ανάγκες εκείνων που σωστά θέλουν να διαφυλαχθούν τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τη διαδικασία, δεν υπήρξε υποστήριξη για την ιδέα άλλου τεχνικού τριμερούς διαλόγου. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν σπατάλι χρόνο. Πρώτερες εμπειρίες το έχουν δείξει. Και ότι αυξάνεται η σύγχυση με αυτού του είδους τους ε, διαλόγους και δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Εγώ στηρίζω την επιθυμία της Επιτροπής να προχωρήσουμε προς επίσημο διάλογο για να ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία ή δυνατόν. Κυρία Γκουρμάη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη παπουσίας αλλά είχαμε ψηφοφορία σε άλλες επιτροπές. Άκουσα τις πληροφορίες από τους συναδέλφους όμως. Έχουν μειωθεί τα χρονικά περιθώρια για τη διεκπαιρέωση υποθέσεως πριν τη λήξη της θητείας. Έχουμε πίεση. Όμως έχουμε πλησιάσει περισσότερο από ποτέ στο θεσμικό αυτό κεφάλαιο και υπάρχει και η απέτηση των πολιτών να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα. Και το τελευταίο σημείο που απειληθεί τάχιστα, ίσω σε ένα τεχνικό τριμερή διάλογο αυτή την εβδομάδα, ίσω την Πέμπτη από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θα ήταν σημαντικό βήμα. Βεβαίω όμω θα πρέπει να παραμείνει όλη η ορμή. Έχουμε καταβάλει πολλέ προσπάθειε και είναι κρίμα να σταματήσουμε τώρα που υπάρχει δυνατότητα συμφωνία. Και αυτό θα ήθελα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί πάση θυσία. Ξέρετε ότι είμαι πρακτική και ρεαλίστρια. Πρέπει να κάνουμε περισσότερους συμβιβασμούς, είναι σαφές. Το Συμβούλιο όμως θα πρέπει να έρθει στα μισά του δρόμου και να μας συναντήσει σε κάποια σημεία. Η υιοθέτηση του νομικού καθεστώτος είναι κρισίμου σημασίας, αλλά όχι αν σημαίνει την έγκριση μιας προτάσεως καινής περιεχομένου. Χρειαζόμαστε να συνεργαστούμε και να καταρτήσουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο και παρατείνω το Συμβούλιο να μας δει την τελική εκδοχή του εγγράφου εργασίας και τα σημεία που φαίνεται στα οποία συμφωνούν αντιπροσωπείες. Αν υπάρχει κείμενο είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψει κανείς. Διαφορετικά θα καταλήξουμε ξανά με έγγραφα της τελευταίας στιγμής και ελάχιστο χρόνο για συζήτηση στη διαπραγματευτική ομάδα και συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο. Μιλώ για συνομιλίες Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πολιτικά ζητήματα. Για την ενιαία αρχή πρέπει να υπάρχουν μέτρα διαφύλαξης όπως η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Σοφών που θα πρέπει να έχει βάρος η άποψη αυτή ακόμα και αν δεν είναι νομικά δεσμευτική. Γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα κάποιο σταυροδρόμι. Μπορεί να χάσουμε όλα όσα προσπαθήσαμε να μαζέψουμε μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αν έχουμε ένα καλό έγγραφο από το Συμβούλιο Εγκαίρος, τότε κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να το διαβάσει και να είναι ενήμερο. Εγώ ε, πιστεύω ότι χρειάζεται και επίσημο τριμερής διάλογος, αλλά χρειάζεται και τεχνικός ε, τριμερής διάλογος για να γίνει κυδαίουσα προετοιμασία. Αυτά και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ ισχύει ακόμα περισσότερο από ότι σε άλλα θέματα ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση του υλικού αντικειμενικού επίπεδου και του επίπεδου που θα χαρακτήριζα ας πούμε διαδικαστικό που αφορά το πόσο έτοιμοι είμαστε να προχωρήσουμε αποτελεσματικά και να βρούμε αποφάσεις. Κάνουμε συνεχώς συζητήσεις ε, επί της ουσίας. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πρόβλημα. Ε, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Περιορίσαμε τον κύκλο των ε, υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων και τώρα αναζητούμε λύσεις που μπορούν να ληφθούν μέσα από τον τρίλογο. Επειδή η διεύθυνση του τριλόγου στο Συμβούλιο δυστυχώς δεν είναι τόσο ευτυχής και επιτυχής εν προκειμένου, είναι σημαντικό πρώτον αυτό που δεν το κατάλαβαν ίσως όλοι ε, στο, ότι Συνδράμουν κι άλλες αντιπροσωπείες ε, στο Συμβούλιο και φροντίζουν από τα παρασκήνια να υπάρξουν συμφωνίες, ενώ δεν είναι παρούσες αυτές ε, ε, ή δεν είναι διαφανείς στο πώς εργάζονται όταν μιλάει η Προεδρία, αλλά νομίζω ότι μπορούμε μέσα από τα λεγόμενα να ακούσουμε πού βρίσκονται οι προεργασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία. Και ακριβώς επειδή το Συμβούλιο εδώ δεν δείχνει μεγάλη συνέπεια ούτε αποτελεσματικότητα στις διαπραγματεύσεις, είναι ακόμα πιο σημαντικό να το κάνουμε εμείς αυτό σωστά και ως Κοινοβούλιο να μην ξαναγυρίζομαι σε θέματα που έχουν ήδη αποφασιστεί ή είναι όριμα προς λήψη απόφασης. Αυτό θα ήθελα να το πω έτσι σαν πρόλογο, εισαγωγικά. Όταν ακούει κανεί την εισηγήτρια, Πολλέ φορέ δεν είχε την εντύπωση ότι έχουμε προχωρήσει τόσο όσο αντικειμενικά έχουμε προχωρήσει. Την τελευταία φορά που συνεδριάσαμε για να προετοιμάσουμε τον τρίλογο, αυτό που είπαν οι συντονιστέ των ομάδων ήταν πολύ πιο προχωρημένο και επικοδομητικό και σαφέ από αυτό που κατέληξε τελικά στα αυτιά του Συμβουλίου. Οπότε πρέπει να προσέξουμε την παρουσία μας, τι παρουσία θα έχουμε ούτως ώστε να μην συμβάλλουμε και εμείς στο να κινούμεθα σε κύκλους συνέχεια στον τριλόγο. Επί της ουσίας νομίζω ότι θα πρέπει με την ανεξάρτητη αρχή ε, ε, υπό το κοινοβούλιο να έχουμε μια κατεύθυνση της διαδικασίας και καθοδήγηση της διαδικασίας που ε, θα είναι από αποπολιτικοποιημένη, αποκομματικοποιημένη και δεν θα έγινε και θα φέρεται από τις πολιτικές ομάδες, αλλά θα είναι θεματοφύλακας του δικαίου που δημιουργήσαμε με βάση τον εσωτερικό κανονισμό και θα διαχειρίζεται τη διαδικασία. Αυτό ισχύει και για την εγγραφή και θα ισχύει και για τη διαγραφή. Το Κοινοβούλιο εδώ παίζει σημαντικό ρόλο γιατί μπορεί να ε, ε, εκφέρει αντίρρηση στην απόφαση, αλλά δεν θα ε, ψηφίζουμε αν θα διαγραφεί μια, ομα... μια... ένα κόμμα ή όχι. Αυτό είναι καλή απόφαση. Δεν θέλω να θυμίσω αυτά που συζητήσαμε ξανά και ξανά, ότι δεν πρέπει να αναλάβει το ρόλο το Κοινοβούλιο να είναι ο ίδιος ο φορέας της λήψης των αποφάσεων, αλλά θα συμμετέχει έντονα στις αποφάσεις. Αλλά δεν θα το αναγάγουμε αυτό σε μια πολιτική απόφαση, όπως και αν εννοούμε αυτήν κάθε φορά. Αλλά θα το κάνουμε μια απόφαση με βάση του δικαίου, όπου θα ασκεί τον σημαντικό του ρόλο το Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι εμείς μπορούμε να λάβουμε απόφαση για αυτούς ε, που μένουν να κάνουν ένα μικρό βήμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουν. Δεν ξέρω πόσο ακόμα θα ε, γυρίζουμε σε κύκλους και δεν ξέρω τεχνικός τρίλογο τι δουλειά έχει εδώ πέρα. Εμεί φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να λάβουμε μια πολιτική απόφαση. Ρώτησα προηγουμένω κατά πόσο υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια για την εγγραφή και τη χρηματοδότηση. Το κείμενο αναφέρει την απέτηση για τουλάχιστον ένα από τα μέλη τους να είναι ευρωβουλευτής αλλά μόνο αναφέρει αυτό το θέμα στα, στα πλαίσια της σηματοδότησης. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω είναι και προϋπόθεση για εγγραφή. Αν περί αυτού πρόκειται, ποιο είναι το μειονέκτημα ένα κόμμα να μην είναι εγγεγραμμένο εν συγκρίση με να είναι εγγεγραμμένο αλλά μην χρηματοδοτείται. Κύριε Πρόεδρε, προτείνατε νομίζω η απόφαση περί να βασίζεται επί κοινοβουλευτικής ε, ψηφοφορίας. Όμως το θέμα των πολιτικών αξιών δεν είναι αντικειμενικό κριτήριο. Το να κρίνει κανείς κατά πόσο ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση είναι δημοκρατικό ή μη δημοκρατικό είναι κάτι υποκειμενικό σαν κριτήριο. Εγώ θα έκρινα πολλές κυβερνήσεις κρατών μελών σαν μη δημοκρατικές όσον αφορά την προσέγγιση τους στην νομοθεσία. Ίσως διαφωνείτε μαζί μου. Η ιδέα ότι η πλειοψηφία των πολιτικών στη, στο Κοινοβούλιο θα έχει δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις για τη μοίρα μιας μειοψηφίας πολιτικών είναι σαφώς και αυταπόδεικτα εσφαλμένο. Εγώ είμαι αντίθετο στην ιδέα της χρηματοδοτήσεως ή ουδήποτε κόμματος. Τα κόμματα θα πρέπει να είναι αρκετά δημοφιλή για να αυτοχρηματοδοτούνται. Αν όλα τα κόμματα ελάμβαναν χρηματοδότηση και εγγραφή θα ήταν μη σοφή χρήση δημοσίων πόρων, αλλά το έστω θα ήταν τίμια τέτοια χρήση. Αν κάποια χρηματοδοτούνται και κάποια όχι, τότε αυτό δεν είναι απλώς κάτι μη σοφόν αλλά διεφθαρμένη χρήση των δημοσίων χρημάτων. Ευχαριστώ. Καλώς. Πρέπει να συνεργάγω συμπεράσματα. Σίγουρα διαφαίνεται ότι υπάρχει μία επιθυμία για να οργανωθεί επίσημος πολιτικός τριμερής διάλογος σύντομα. Δεν νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίσουμε τους τεχνικούς να συναντηθούν αν επιθυμούν κάτι τέτοιο άτυπα. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό θα ήταν κάτι χρήσιμο για να βοηθήσουν, να προετοιμάσουν όπως είπε και η κυρία Γκουρμάη. Ε, ε, εφόσον λοιπόν αυτή η άποψη τριμερούς διαλόγου τεχνικής φύσεως αυτή την εβδομάδα προέρχεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ λέω αν θέλουν να το κάνουν, να το κάνουν. Εμείς από την πλευρά μας ζητούμε να λάβει χώρα πολιτικός τριμερής διάλογος ταχύτερο δυνατόν, να καταλήξει συμπεράσματα και θέλουμε να γίνει άλλη μια συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων και τεχνικών εμπειρογνωμόνων να λάβουν υπόψη το επίπεδο στο οποίο φτάσαμε και να προτείνουν λύσεις, πώς να το πω, που επιτρέπουν ε, στη, από την ψηφοφορία την επιλογή ε, σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό είναι το πιο υγιές. Αν θέλουν να το κάνουν, ας το κάνουμε. Το κάνουμε κατά το παρελθόν συνεδρία σε τρεις ομάδες, οι τρεις νομικές υπηρεσίες και τι μας Αυτό δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε. Επίσημα όμως θα ζητήσουμε να διεξαχθεί πολιτικός τριμερής διάλογος το ταχύτερο δυνατόν. Συμφωνούμε. Καλώς. Δεν βλέπω διαφωνείς, οπότε ολοκληρώνεται έτσι η συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε την 3η 26 Νοεμβρίου από τις 15-18.30, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου από 1530 έως 18.30 και 3η 17 Δεκεμβρίου από τις 9 ως τις 12.30. Να υπενθυμίσω ότι το απόγευμα υπάρχει ακρόαση, συζήτηση όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών και διάφορες οργανώσεις που προσεκλήθησαν δυνάμει του άρθρου 17 της Συνθήκης Λισαβόνας εκκλησίες και κοσμικές οργανώσεις θα συμμετάσχουν. Υπάρχουν πολλές κοσμικές, περισσότερες οι κοσμικές αυτές οργανώσεις, αυτές θρησκευτικέ, αλλά αυτή θα είναι χρησιμότατη συνάντηση για να δούμε τις οργανωμένες εκφάνσεις κοινωνίας των πολιτών Λοιπόν, θα σας έλεγα να είσαστε παρόντες απόψε από τις 3 το απόγευμα εδώ, σε αυτή την ακρόαση. Ευχαριστώ. Γεια σας.